και ιδιαίτερα στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα τα οποία έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Thank you, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έκθεση Κλίντς δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας. Ο λόγος στον εισηγητή. Τέσσερα λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αν ξεπεράσω τα τέσσερα λεπτά, νομίζω έχω άλλα δύο, οπότε ενδεχομένως θα πάρω όλο το χρόνο ομιλία για να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Η αρχική πρόταση του 2003 ήδη από τότε ήταν αντικείμενο κάποιων τροποποιήσεων. Το 2009, το Σεπτέμβριο, ξεκίνησε η επεξεργασία αυτών των νέων ε, προτάσεων όσον αφορά τις κινητές αξίες και τις απαραίτητες ρυθμίσεις στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Η σημερινή αναθεώρηση, αν θέλετε, έχει κάποιες τεχνικές πτυχές και ανταποκρίνεται στα σημερινά νέα δεδομένα των χρηματαγορών. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, σκιώδες εισηγητές και άλλους, οι οποίοι με βοήθησαν. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και δεν θα ήταν δυνατόν σε λιγότερο από 10 μήνες να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που φτάσαμε με αυτό το πακέτο προτάσεων, εάν δεν υπήρχε αυτή η εξαιρετική συνεργασία. Όσον αφορά τον τρίλογο, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν οκτώ σημεία στα οποία μπορούμε να βρούμε συμφωνία. Καταρχήν, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πρόσβαση στο κεφάλαιο, ο σκοπός των προτάσεων μας είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μπορούν δηλαδή να χρηματοδοτηθούν από τις χρηματαγορές και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη δυνατότητα για τις μικρές επιχειρήσεις, κάτι που μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατον. Κάναμε λοιπόν κάποιες αλλαγές που θα διευκολύνουν στην την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέσαμε δε ένα ανώτατο όριο το οποίο είναι των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η διευκόλυνση είναι κάτι που θα πρέπει να είναι χρήσιμη για όλες τις μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα γιατί ανεβάσαμε το όριο των 50.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ. Όσον αφορά την δομή του κεφαλαίου, του μετοχικού κεφαλαίου αυτών των επιχειρήσεων, είδαμε για άλλη μια φορά τις προϋποθέσεις και τους όρους που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, προσφέροντας νέες προοπτικές ε, για τους συνεργάτες αυτών των εταιριών και πάλι προσπαθώντας να μειώσουμε το διοικητικό και γραφειοκρατικό άχθος, δίνοντας πληροφορίες σε όλους τους συνεργάτες αυτών των επιχειρήσεων που επιθυμούν να καταρτιστούν. Διασφαλίσαμε δε κάποιες εταιρείες οι οποίες ε, βρίσκονται στην, ε, στα χρηματιστήρια ενός άλλου ευρωπαϊκού κράτους να μπορούν να προσφέρουν στους εργαζόμενους τους που βρίσκονται σε μια άλλη χώρα τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αυτές τις νέες διατάξεις και από τις κινητές αξίες. Τώρα, Περιληπτικά θα ήθελα να πω ότι δεν απαιτώ από όλους να διαβάσουν τις πολυάριθμες σελίδες αυτού του σχεδίου. Έχουμε μια συνοπτική έκδοση με τις βασικές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για έναν επενδυτή που θέλει να επενδύσει με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι σε αυτό το συνοπτικό έγγραφο πραγματικά υπάρχουν οι πληροφορίες κλειδιά και συμφωνήσαμε σε αυτήν την συνοπτική έκδοση να εξετάσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όντως οι ουσιαστικές, οι κύριες πληροφορίες είναι παρούσες και θέλουμε να περιορίσουμε το έγγραφο αυτό σε 20-30 σελίδες, να είναι δηλαδή ένα κείμενο ευανάγνωστο, έτσι ώστε ο απλός ε, επενδυτής να μην χάνεται. Έχετε 4 συν 2 λεπτά. Πολύ περιληπτικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, τελειώνω. Όσον αφορά την αστική ευθύνη, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια νέα πρόταση για τον μεσολαβητή, τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτής της μεσολάβησης, υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για τις διάφορες διαδικασίες. Έβδομο σημείο, η ρήτρα αναθεώρησης, πέντε χρόνια αυτό το έγγραφο, αυτή η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί μετά από πέντε χρόνια. Έχω πολύ σύντομα το 8ο και πολύ σημαντικό σημείο, το τελευταίο σημείο, το πρώτο έγγραφο που ουσιαστικά συμμορφώνεται και συμβαδίζει με την Λισαβόνα. Προσπαθούμε εδώ να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει αρκετό χρόνο. Είχαμε τρεις μήνες για να αντιδράσουμε στις προτάσεις της Επιτροπής. Ζητούμε άλλες τρεις μήνες και πραγματικά θα θέλαμε να ξέρουμε αν μπορεί να δοθεί η λεγόμενη πρόορη ε, έγκριση, early approval, για το κείμενο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όταν στις 13 Ιανουαρίου πέρασα από την ακρόαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν διοριστώ ως επίτροπος, ε, ε, υποσχέθηκα ότι θα προστατεύσω τους επενδυτές και ότι θα περιορίσουμε το γραφειοκρατικό άχθος το οποίο υφίσταται οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το βασικό κομμάτι του οικονομικού ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτή η οδηγία που, διευκολ... που απλουστεύει ε, τις συναλλαγές για τις κινητικές αξίες που διευκολύνει το έργο των μικρών, μικρο, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τις διευκολύνει να έχουν πρόσβαση ε, στις κεφαλαιογορές, ε, για μας αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα και πιστεύουμε ότι ε, η συνεισφορά του Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ σημαντική και το Συμβούλιο αλλά και η Κομισιό έπαιξαν το ρόλο τους και εξ ονόματος της Κομισιό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Πλίνσε και την Οικονομική Επιτροπή. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα με αυτό το κείμενο του συμβιβασμού που έχουμε στα χέρια μας και που βελτιώνει το αρχικό πνεύμα, αν θέλετε, της πρότασης. Η οδηγία του 2003 είχε έναν πολύ καλό στόχο, τον οποίο και εξυπηρέτηση, για τις ε, σαφείς οδηγίες που έπρεπε να ακολουθούν όσοι εξέδιδαν κινητές αξίες και και το προσπέκτους αυτό ε, ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το προσπέκτους του 2003 πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε την ε, νομική διαφάνεια του κειμένου. Και χάρη σε εσά και χάρη στην αναθεώρηση που έγιναν, κάποιες, κινητε, κάποιες εκδόσεις κινητών αξιών θα πρέπει να σέβονται το την υποχρέωση δήλωσης ε, ούτως ή άλλως ε, η μορφή και η παρουσίαση του προσπέκτου θα βελτιωθούν σε περίπτωση που οι εταιρείε ε, κάνουν πωλήσει χρησιμοποιώντας μεσολαβητές ή που διανέμουν μετοχές τους εργαζομένους τους. Και θα πρέπει ε, να καταργήσουμε και τις διατάξεις ε, που ε, επικαλύπτονται με, τις, με υπάρχουσες οδηγίες. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η νέα αυτή πρόταση αποτελεί μια προσαρμοσμένη απάντηση στις ανάγκες ε, των φορέων της αγοράς είτε πρόκειται για αυτούς που εκδίδουν και τις αξίες είτε για αυτούς που τις αγοράζουν. Ε, η Κομισιόν σέβεται επομένως στις υποσχέσεις της για μεγαλύτερη διαφάνεια, για περιορισμό της γραφειοκρατίας και ανεβάζοντας το επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Πραγματικά πρόκειται για μια δυναμική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οποία την ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ο επόμενος ο, θα έπρεπε να ήταν ο κύριος Μπόντου, που δεν είναι εδώ όμως, δεν τον βλέπω. Ο κύριος Φέιο έχει το λόγο τώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά. Είχαμε πολύ καλές προτάσεις από τα μέλη και θα ήθελα να υπογραμμίσω τον θετικό ρόλο του κ. Κλίντς προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Μιλώντα για ενημερωτικά φυλάδια, μιλάμε ασφαλώς για την ιδέα της ε, δημοσίευσης στοιχείων της σιγουριάς σε μια αγορά και της καλύτερης ε, πρόσβασης σε επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο μερικές ε, φορές υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και την προστασία των επενδυτών που και οι δύο είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήγουμε σε ε, ισορροπία και αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε αυτή την αναθεώρηση δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σκεφτήκαμε ιδιαίτερα την ανάγκη να σεβαστούμε τους μικρούς επενδυτές. Προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη απλο... απλοποίηση, μικρότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τα πολλές φορές υπερβολικά διοικητικά βάρη. Στον τριμερή διάλογο δεν πήγαμε με οι τσίρες απόψε ο καθένας, αλλά καταφέραμε και βρήκαμε μια ισορροπία. Νομίζω ότι με αυτό το κείμενο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σιγουριά σε ευρωπαϊκές αγορές στο μέλλον. Ο λόγος στον κύριο, στην κυρία Στήλερ, συγγνώμη, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, thank you, Mr. President, and... Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους κοιόδους εισηγητές για τη συνεργασία τους. Πιστεύω ότι επετεύθη ένα συμβιβασμός και έγινε δεκτός ο συμβιβασμός αυτός γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ε, προστασία για τους επενδυτές, κυρίως για τους μικρομεσαίους επενδυτές που ούτως ή άλλως και αυτό ήταν και το πνεύμα της αρχικής ε, οδηγίας όπως είπε και ο Επίτροπος. Εάν δούμε ε, και όπως είπε και ο κύριος Κλίνς τι θέλαμε ήταν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και θέλουμε την ευθύνη να την έχουν οι, οι βασικοί επενδυτές. Διευκρινίσαμε επίσης ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την, το ποιον, ποιο, την, την, ποιος είναι υπεύθυνο σε περίπτωση κυρίως που υπάρχει και ένας διαμεσολαβητής και δεν είναι απευθείας η συναλλαγή ανάμεσα στον εκδότη και στον, στον αγοραστή. Πιστεύω ότι είναι ευπρόσδεκτο το βήμα που έγινε να, να ορίσουμε ποιος, ε, ποια είναι καταρχάς ε, η αντιμετώπιση μιας τρίτης χώρας, ε, αυτός ο επενδυτή ο οποίος έχει περισσότερα προσόντα από αυτά τα οποία χρειάζονται και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να επενδύσουν στην εταιρεία τους, μήπως οι εργοδότες θα πρέπει να το λάβουν αυτό ε, υπόψη τους. Εγώ θα χρησιμοποιούσα την οδηγία για το προσπέκτους σαν, ε, μία, σαν ένα ορόσημο. Όσον αφορά την δημοσίευση του προσπέκτους που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή όχι, αυτό είναι ευπρόζεκτο νομίζω, όπως επίσης και αναθεώρηση ανά πενταετία. Επομένως, σε γενικές γραμμές ε, η οχι αυτο ειναι ευπροζεκτο νομιζω οπως επισης και να ανα αναπενταετία. επομενως σε γενικες γραμμες η ομαδα μας ε, δέχεται την ε, συμβιβαστική πρόταση την οποία καταλήξαμε και θα υποστηρίξουμε το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμίτ για τους ε, φιλελεύθερους για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν της χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, και υπό το φως της ε, χρειάζεται μια καλύτερη ρύθμιση των αγορών. Αλλά κυρίως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία. Και πιστεύω ότι δεν θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία αν δεν ε, έχουμε ένα σύστημα ισορροπημένο, ένα σύστημα προστασίας ισορροπημένο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κλίντς γιατί δούλεψε πολύ καλά ε, αντιδρώντας σε μια υπερβολικά λεπτομερή νομοθεσία. Ε, διαγράφηκαν και καταργήθηκαν όλες οι περιττές υποχρεώσεις που θα βάρεναν τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κλίντς μαζί με τους συναδέλφους και μαζί με την ε, ομάδα μας ε, δουλέψαμε, ε, δούλεψε, δουλέψαμε όλοι μαζί και είμαστε ικανοποιημένοι διότι αυτή τη στιγμή πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βαρύνονται από υπερβολικές διοικητικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι έτσι διευκολύνεται και ο ρόλος των επενδυτών. Μιλήσαμε για, τις, για τα κατόφλια των καινούριων εκδόσεων και νομίζω ότι οι ε, προτάσεις που επελέχθηκαν ε, είναι ισορροπημένες. Τα κατόφλια θα πρέπει να την χάνουν σεβασμού και να εφαρμόζονται ακριβώς για να αποφασίσουμε αν θα εκδίδεται ή όχι ε, ενημερωτικό δελτίο. Και στη σχέση με τις τρίτες χώρες ε, έχουμε πολύ ισορροπημένα κατόφλια. Συνοψίζοντας, όπως είπε και η συνάδελφος ε, του σοσιαλιστικού, σοσιαλιστικής ομάδας, θέλω και εγώ να, συν, να συγχαρώ τον κύριο Κλίντς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα γιατί θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την κατάσταση εκατομμυρίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η κυρία Ford για τους ιδρυτικούς μεταρρυθμιστές. Um, Commissioner... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι ίσως μία από τις πιο συναρπαστικές εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε, γιατί ουσιαστικά παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την ρύθμιση των, ε, της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις κεφαλαίες αγορές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και ήταν εξαιρετική συνεργασία σαν σκιώδης εισηγήτρια με τον εισηγητή, τον κύριο Κλίντς και πραγματικά η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου μας οδήγησε μετά από την συνεργασία που είχαμε σε ένα ευανάγνωστο κείμενο, σε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις ε, χρηματαγορές. Σαφώς και θα χρειαστούν κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους επενδυτές και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στο συνοπτικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες, τις πιο σημαντικές τις πληροφορίες κλειδιά. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρές. Σε μια εποχή όπου οι αγορές κυμαίνονται με έναν τρόπο που δεν μπορεί να ελεγχθεί, θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε αυτή την πρόσβαση στις χρηματαγορές. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα φανούν οι επιπτώσεις αυτής της πρότασης. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου και οι επενδυτές αλλά και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν από ένα συγκεκριμένο μέτρο που πήραμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκαρσία, ο κύριος Γκαρσία. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Ξέρουμε διάφορα πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η κρίση ήταν σαν, ε, μια μεταλλα, σαν ένα μεταλλασσόμενο ιό. Ήταν δημοσιονομική, μετά έγινε τραπεζική, μετά έγινε οικονομική και μετά έγινε κρίση δημοσίου χρέους που μπορεί να προκαλέσει και άλλη κρίση με τη σειρά της. Ξέρουμε επίση ότι κόστησε πολύ ακριβά. Σύμφωνα με τι δικέ υπηρεσίε, οι ενισχύσει που έχουν προβλεφθεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα φτάνουν τα 3,53 εκατομμύρια δολάρια. Το 1 τρίτο δηλαδή του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης γνωρίζουμε ότι ένας από, μία από τις αιτίες της κρίσης ήταν η έλλειψη διαφάνειας σε προϊόντα, ε, όργανα και αγορές. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντική η έκθεση την οποία συζητούμε. Αν να σας υπενθυμίσω επίσης ότι μόνο στις ΗΠΑ την περιοδο 2000-2006 τα τέτραπλασιάστηκαν ε, τα, τετραπλασιάστηκε το ποσό το οποίο ε, κυκλοφορούσε ως κινητές αξίες. Ε, μάλιστα υπήρχαν τράπεζες που δηλώσαν ότι δεν ήξεραν τι πουλούσαν. Επίσης γνωρίζουμε ότι πολλές από τις υποσχέσεις που δώσαμε στο G20 και τις δεσμές που αναλάβαμε δεν ξεπέρασαν τη σφαίρα της φαντασίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι στην αναμόρφωση του, του χρηματοπιστικού συστήματος πρέπει να ξεκασφαλίσουμε τα εξής τρία. Οι, ε, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, τα ευρωπαϊκά ιδρύματα θα πρέπει να την χάνουν ε, ελέγχου από ευρωπαϊκά όργανα. Δεύτερον, θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου ουσιού στο μέλλον. Και τρίτον, οι ασθένειες οποίες δεν έχουν προκληθεί από τους ε, πολίτες μας, θα πρέπει να αποφύγουμε λέω, αυτές οι ασθένειες να πληρώνονται από τους ίδιους πολίτες. Δεν ε, θέλουμε να ευνηδιαστούμε από την επόμενη κρίση. Και θα ήθελα πάντοτε να σας ευχηθώ τόλμη, τόλμη, τόλμη στα καθήκοντά σας κύριε Επιτροπέ. Μαγκάγιο, τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Κούτας για ένα λεπτό suprimarea ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η διπλή διαφάνεια, η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις ε, χρηματαγορές, σαφώς και θα μας οδηγήσει σε μια σημαντική εξοικονόμηση των 173 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και βλέπουμε ότι μέχρι το 2008 το 2002 πολλές τέτοιες επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το χρέος οφείλεται πολλές φορές στο διοικητικό και το γραφειοκρατικό βάρος το οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις αυτές. Ο συντονισμός είναι απαραίτητος μεταξύ των κρατών μελών και αυτό ισχύει και για το έγγραφο. Ο κύριος Κάζα, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Είδαμε πολλές αναταραχές τα τελευταία χρόνια και πολλοί έχουν πληγεί. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές, κυρίως οι μικροεπενδυτές, θα τύχουν της απαραίτητης προστασίας στην Ευρώπη, ότι θα έχουν τις πληροφορίες για να μπορούν να παίρνουν εν επιγνώση τους τις αποφάσεις που θέλουν να πάρουν για να επενδύσουν. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ασφάλεια στις ευρωπαϊκές αγορές για να προσελκύσει νέους επενδυτές. Θα πρέπει να υπάρξουν και να επικρατήσουν ευρωπαϊκά πρότυπα όπως ακριβώς έγινε και με την ε, οδηγία UCITS. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να προσαρμόζονται και να αναθεωρούνται. Συμφωνώ απολύτως ότι κάποιες από αυτές τις προτάσεις δεν είναι χρήσιμες και ότι θα πρέπει να μην αναγράφεται ο αριθμός αυτών οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφώνονται. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθεί ένα σημαντικό βάρος και εμπόδιο για τις επιχειρήσεις. Τα κράτη-μέρη θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν αυτά τα κοινά πρότυπα. Κυρία Πρόεδρε, τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κλέτς, τον εισηγητή, για την εξαιρετική του έκθεση και τους σκιώδες εισηγητές επίσης, γιατί θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι ισορροπημένη και επίκαιρη. Τώρα η κυρία Σάγια για δύο λεπτά. puhemies. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι η έκθεση για την τροποποίηση της οδηγίας είναι πάρα πολύ καλή. Μειώνουμε το διοικητικό άχθος και ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές έκαναν πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι η προστασία των επενδυτών θα πρέπει πάντοτε να είναι στο μυαλό μας. Η νομική βεβαιότητα ε, αυξάνεται με αυτό το κείμενο, βελτιώνεται και η νομική βάση έχει πλέον περιοριστεί. Τα ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να συντάσσονται εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται αντιφάσεις και παραπλανήσεις. Πιστεύω ότι αυτή η ενότητα του μορφοτύπου των ενημερωτικών δελτίων τα κάνει πιο ευανάγνωστα. Έχω υποβάλει μία τροπολογία έτσι ώστε όλοι οι επενδυτές να τη χάνουν της ίδιας και ίσης μεταχείρισης. Δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε. Πολλές φορές οι μικροί επενδυτές γνωρίζουν λιγότερα από τους μεγαλύτερους επενδυτές. Και σκοπεύω να το επαναλάβω αυτό και στο μέλλον. Η οδηγία έχει ένα σημαντικό στόχο. Ο επενδυτής θα πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση σαφής διαθέσιμες πληροφορίες. Νομίζω ότι η τροποποιημένη οδηγία θα συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάγια. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο ο, τρεις συνάδελφοι. Σας παρακαλώ πολύ να κρατήσετε το χρόνο του ενός λεπτού στην κάθε παρέμβαση. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Κύριε θα Κύριε Κλίντ, σας ευχαριστούμε πολύ για την εργασία σας και θα ήθελα να πω το εξή. Η, πρόταση της Κομισιόν να διευκολύνει την δημοσίευση αυτού του έγκυρου ενημερωτικού δελτίου ε, βοηθάει τους ε, επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους ε, τις κατάλληλες και αναγκαίες πληροφορίες και αυτή η ενημέρωση ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή αγορά αν θέλετε. Πρέπει να έχουμε επομένως ένα σαφές νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες και βεβαιότητες όσον αφορά την ε, αξιοπιστία του κράτους υποδοχής. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε επίσης να περιορίσουμε και το κόστος και το γραφειοκρατικό άχθος μέχρι το 2012. Επίσης ήθελα να αναφέρω ότι οι νέες διατάξεις θα προστατεύσουν καλύτερα τους επενδυτές δίνοντάς τους την ευκαιρία ευκαιρία να αναλύουν καλύτερα τους κινδύνους που έχουν οι κινητές αξίες πριν προχωρήσουν στην επένδυσή τους. Το λόγο θα πάρει ο κύριος Σόμπερ Μάγερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι κεντρικές αρχές σαφώς και χρειάζονται μια ενιαία ρύθμιση όσον αφορά τις κινητές αξίες για να προστατεύσουμε τους επενδυτές. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση αυτών των ε, επενδυτών θα πρέπει να ακολουθείτε με απαραίτητη πληροφόρηση. Πληροφόρηση η οποία θα έρχεται σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν αυτό που καλούνται να κάνουν γνωρίζοντας τις πραγματικές αξίες. Το θέμα της ευθύνης, της αστικής ευθύνης όπως ξέρετε εξαρτάται από τη νομική κατάσταση που είναι τελείως διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη. Θέλουμε λοιπόν διαδικασίες με διαφάνεια, κάτι το οποίο να ξεπερνάει αυτές τις διαφορές. Η νομική βάση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρε η κυρία Βερτμάνα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, το ενημερωτικό δελτίο αυτό αναφέρεται στις ε, σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει ένας επενδυτής ο οποίος θέλει να έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές. Όσον αφορά τη διαφάνεια, όσον αφορά τους ελέγχους, θεωρώ πολύ θετικό βήμα αυτό που γίνεται σήμερα για την προστασία των μικρών επενδυτών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σαφώς και θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση, πιο εύκολη για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις στο μέλλον. Είσαστε και πολύ σύντομοι στον χρόνο. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μπαρνιέ, εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ένα προς ένα τους ε, ομιλητές, γιατί βλέπω ότι εγκρίνουν, επιδοκιμάζουν το κείμενο αυτό, το οποίο είναι ένα κείμενο συμβιβασμού, είναι ένα δυναμικό κείμενο, κείμενο το οποίο δεν θα μπορούσε να ε, συμπεριλάβει όλες τις προτάσεις που είχαν γίνει, αλλά πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο, ε, ο κ. Κλίντς, η Επιτροπή Τζούρι κλπ. έχουν λόγους να είναι ικανοποιημένοι. Γιατί, Γιατί το κείμενο έχει ωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα σχόλιά σας και από την επικοδομητική κριτική την οποία εκφράσατε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ένας μεγάλος αριθμός ε, τροπολογιών υποβλήθηκε από εσά και υιοθετήθηκε. Το πεδίο εφαρμογής, διατάξεις ε, για τις ε, πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου, η λησβονοποίηση, να το πούμε έτσι, του κειμένου κλπ. Ο κ. Φέιο αναφέρθηκε στην σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των επενδυτών και στην προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ε, το ενημερωτικό δελτίο θα, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι προσαρμοσμένο ε, έτσι ώστε να μην αποτελεί ιδιαίτερο αχθός. Τις έχουμε λάβει υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και ταυτόχρονα θα σεβόμαστε και θα προστατεύουμε τους επενδυτές. Ε, ένα άλλο θέμα της κυρία Σισάγια. για τους ε, επενδυτές και τους ιδιώτες. Η οδηγία λαμβάνει υπόψη ε, τη διαφορά ανάμεσα στους δύο προκειμένου να εξασφαλίσει την επαρκή προστασία των ιδιωτών. Η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί όλες τις ε, τροπολογίες και υποστηρίζει το κείμενο. Όπως το υποστήριξαν οι ομιλητές και ο εισηγητής. Νομίζω ότι το κείμενο είναι ένας καλός συμβασμός και είμαστε σίγουροι ότι η οδηγία θα κάνει τη διαφορά στην προστασία των επενδυτών και στην μείωση των διοικητικών βαρών για τους εκδότες. Θα ε, επιτρέψει να δημιουργήσουμε πραγματική αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκαρσία Μαργκάγιο για αυτά που είπε, γιατί πέραν του κειμένου, το οποίο αποτελεί πρόοδο, ε, ενέγραψε ο κ. Μαργκάγιο την πρόοδο αυτή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο εργάζεται ο ίδιος, στο πακέτο επιτήρησης. Είναι το πλαίσιο της διαφάνειας. Νομίζω ότι με το κείμενό μας βελτιώνουμε την διαφάνεια, την προσαρμόζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους εκδότες, σεβόμενοι τα δικαιώματα των επενδυτών. Συμπεριλαμβάνουμε παρόμοιες διατάξεις και στο πακέτο επιτήρησης, το οποίο αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ο κ. Μαργκάγιο μαζί με άλλους συναδέλφους. Ε, νομίζω ότι η τόλμη μας αφορά όλους, είναι συλλογική τόλμη, την δείξαμε και Νομίζω ότι όλοι μαζί και με το Συμβούλιο θα χαρούμε ιδιαίτερα από την έγκριση αυτού του κειμένου. Ε, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε συμβασμό και σε άλλα κείμενα τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή, τα hedge funds κλπ. Και το μεγάλο project βέβαια της επιτήρησης στην Ευρώπη. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα κείμενα. Ε, για, τα χρειαζόμαστε και για τους 20 αξιολόγηση για τους οποίους μιλούσαν προηγουμένως αλλά και για άλλες πτυχές της ε, διαφάνειας και της ε, οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής ο κύριος Κλίνς, αλλά επειδή έχει περάσει δι το χρόνο του, μόνο μισό λεπτό, ένα λεπτό κύριε Κλίνς, μόνο για να κλείσετε. Έχετε καλύψει τα έξι λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα Καταρχήν ευχαριστώ τον Επίτροπο, ευχαριστώ όλους όσους με πολύ θετικό τρόπο σχολίασαν την συνεργασία μας. Όντως ήταν εξαιρετική και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται πολύ η εργασία μας. Σκοπός μας είναι να μειώσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια και να προστατεύσουμε και τους Ευρωπαίους επενδυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να αναθεωρηθεί πάλι η οδηγία αυτή για να αποφύγουμε καταχρήσεις και να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών. Πιστεύω ότι τα... οι αξίες αυτές, οι οποίες δεν οδηγούν σε μερίσματα και οι αξίες αυτές, οι οποίες απευθύνονται σε επενδυτές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που βρίσκεται η επιχείρηση, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν. Ε, η συζήτηση έληξε εδώ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού